Λοιπόν, καλώς ήρθατε στη συνεδρία της Επιτροπής. Ψηφίσαμε με τη ΛΥΜΠΕ και ΦΑΜ σε κοινή ε, συνεδρίαση και ήταν ένα καλό πακέτο που καταφέραμε να περάσουμε και που νομίζω θα μας οδηγήσει σε καλύτερες καταστάσεις. Προχωρούμε στην ημερήσια διάταξη και πάμε στο σημείο 14 που έχει τίτλο «Η σεξουαλικοποίηση των νέων κοριτσιών». Θα δώσω το λόγο στην κυρία Σκριβλόσκα. Σκριντλεύσκα μάλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η σεξουαλικοποίηση των νέων κοριτσιών δεν είναι ένα νέο φαινόμενο, επουδενή αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει αυξηθεί πρόσφατα αυτό το φαινόμενο και πλήττει όλο και νεότερες κοπέλες. Ε, Συνδέεται με τις τεχνολογικές εξελίξεις και την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωση, στα ΜΜΕ, κυρίως στο διαδίκτυο. Όσον αφορά τα νέα κορίτσια, αυτή η σεξουαλικοποίηση ε, ε, σε τι συνίσταται. Ε, να επιβάλλεις τεχνητή πρώιμη σεξουαλικότητα στα κορίτσια που δεν είναι έτοιμα ακόμα. Πώς γίνεται αυτό. Με την ε, υπεργολική εστίαση στην φυσική ελκυστικότητα. Να κάνεις τα κορίτσια να πιστεύουν ότι η εμφάνισή τους θα, τους, θα τις οδηγήσει στην επιτυχία. Ε, τα νέα κορίτσια που είναι ελεύθερα να φορέσουν θα έπρεπε να είναι ελεύθερα να φορέσουν ό,τι θέλουν, ό,τι τους αρέσει, προσπαθούν να είναι ελκυστικά, ούτω ώστε τα άλλα κορίτσια και όλοι οι άλλοι άνθρωποι να, τους, ε, να τις δέχονται. Άρα αυτό οφείλεται στην κοινωνική πίεση. Η κοινωνική πίεση τις κάνει να πιστεύουν ότι αυτό αναμένεται από αυτές. Μπορούμε να μιλήσουμε εδώ για τεχνικές μορφές για την εμφάνιση. Αδύνατες όμορφες γυναίκες που τονίζουν τα χαρακτηριστικά τους για να προσελκύσουν τους άντρες. Ε, διασημότητες, επίσης είναι μια συνιστόσα της εικόνας. Οι διασημότητες παρουσιάζονται σαν σύμβολα του σεξ και συνεχώς έτσι τονίζεται το γεγονός ότι είναι ελκυστικά πρόσωπα. Τα περιοδικά δείχνουν κορίτσια σε προκλητικές πόζες και αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο όλα αυτά τα περιεχόμενα είναι κατανόητα για τα κορίτσια που δεν είναι έτοιμα να τα αφομοιώσουν και πέφτουν θύμα σε καταχρήσεις. Και στα σχολεία αλλά και σε άλλα περιβάλλοντα. Η πορνογραφία διαδίδεται όλο και περισσότερο. Ε, υπάρχουν και άλλες συνέπειες όπως διαταραχές ε, διατροφικές, ε, βουλημία, ε, ανορεξία, κατάθλιψη κλπ η συνέπεια της σεξουαλικοποίησης επηρεάζει τα νέα κορίτσια και έχει και μακροπρόθεσμες συνέπειες σύμφωνα με αυτά που λένε οι ψυχολόγοι. Στα ΜΜΕ οι γυναίκες ε, παρουσιάζονται σαν αντικείμενα. Αντικείμενα κατώτερα από τους άντρες και σαν όντα που ο μόνος λόγος ύπαρξής τους είναι η ικανοποίηση των αναγκών των ανδρών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα διακρίσει κατά των γυναικών και στο τόπο εργασία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε μία φωνή, να έχουμε μία στάση κατά της σεξουαλικοποίησης αυτής για να προστατεύσουμε τα νέα κορίτσια και να μειώσουμε τα αρνητικά φαινόμενα στα οποία εκτίθενται οι νέες κοπέλες. Στην έκθεσή μου εστιάζομαι στην ηλικία 6 με 13. Τα κορίτσια πάνω από αυτή την ηλικία είναι ήδη στην εφηβεία και το εύρος ποικίλει από τα 13 μέχρι τα 18. Τονίζουν οι εμπειρογνώμονες, εκεί δεν μπορούμε να έχουμε ενοποιημένα ενιαία πρότυπα. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, από την, ε, μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας δεν μπορεί να ξεπεράσει έναν αριθμό σελίδων και γραμμάτων και λέξεων. Ε, άρα έπρεπε να στεστώ επί των σημαντικότερων θεμάτων. Δεν περιέγραψα τη σεξουαλικότητα και τα αποτελέσματα της σεξουαλικοποίησης λεπτομερώς. Εστιάζομαι στις τάσεις για σχολεία, ιδρύματα, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ ε, και ποιε είναι οι καλές πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, αλλά και πιο πρόσφατα στην Ιρλανδία. Αυτές οι χώρες ανέλαβαν δράσεις κατά της σεξουαλικοποίηση και των αρνητικών της συνεπειών. Όχι μόνο οι κυβερνητικοί φορείς, αλλά και η βιομηχανία, η κλωστοϊφαντουργία και ο διαφημιστικός τομέας ανταποκρίθηκαν θετικά και πρότειναν αυτορύθμιση αυτό σημαίνει ότι γνωρίζει και ο τομέας και η βιομηχανία το φαινόμενο, παρόλο που και αυτοί εν μέρη συμβάλλουν στη διαμόρφωση των κινδύνων που επηρεάζουν και τα νέα κορίτσια αλλά και τα αγόρια. Όσον αφορά το περιεχόμενο της εκθέσεως, θα αναφερθώ στο ρόλο των γονέων. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν περισσότερες δυνατότητες, θα πρέπει να μπορούν να ελέγχουν καλύτερα την πρόσβαση των παιδιών τους στο διαδίκτυο θα πρέπει να μπορούν να προστατεύσουν τα νέα κορίτσια από την κατάχρηση και από τους συνομιλίκους τους και από τους ενήλικες. Παρομοίως όσον αφορά τα παιχνίδια τα ηλεκτρονικά. Χρειάζεται πανευρωπαϊκό σύστημα για τα παιχνίδια. Πρέπει να επεκταθεί το σύστημα για την πληροφορική και να ανακαλύπτει και το σεξουαλικό περιεχόμενο στα παιχνίδια. Και ίσως και το υλικό αν έτσι θα βοηθήσουμε του γονεί προς αυτές τα παιδιά. Ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια για κομπιούτερ το 2008 περιέγραφε την εξή κατάσταση. Οι παίκτε έπρεπε να συνευρεθούν σεξουαλικά με μία πόρνη και μετά έπρεπε να σκοτώσουν το θύμα τους. Και χρειάστηκε παρέμβαση από πολλούς γονείς για να αποσυρθεί το παιχνίδι από την αγορά σήμερα δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Και δεν μπορούν να το αγοράσουν νέα κορίτσια και αγόρια. Στην έκθεσή μου μιλάω και για τους γονείς που άθελά τους, χωρίς να το γνωρίζουν, μετατρέπουν τα παιδιά τους αντικείμενα. Παραδείγματος χάρη μέσω ε, ε, ε, εγχειρήσεων, αισθητικών εγχειρήσεων, επεμβάσεων, ε, όταν βάζουν τα παιδιά του να συμμετέχουν σε καλυστία, Όπω γίνεται στην Ισπανία, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο κλπ. και στι Ηνωμένε Πολιτείε. βέβαια. Αυτοί οι διαγωνισμοί καλονής συμπεριλαμβάνουν διάφορες ηλικιακέ ομάδες και έχουν και μια ομάδα τέτοια ηλικιακή από 0 μέχρι 3 ε, χρόνια, 0 μέχρι 3 ετών. Πολύ συχνά τα κορίτσια πίνουν ε, ποτά με περιεχόμενε θερμίδε για να τονωθούν ενεργειακά, για να μπορούν να παρουσιαστούν καλύτερα στη σκηνή. Στα σχολεία και στα σχολικά μαθήματα θα πρέπει να διδάξουν τα παιδιά πώς να αντιμετωπίσουν το, τα μίδια και το περιεχόμενο των μίδια με κριτική σκέψη. Ε, τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν πώς μπορούν να έχουν καλή οικογενειακή ε, ζωή και το περιεχόμενο στο οποίο εκτίθεται είναι προσαρμοσμένο στην ηλικία τους. Ε, κανονικά θα έπρεπε οι γονεί να ασχολούνται με αυτό το θέμα αποκλειστικά. Αλλά βέβαια έχουν πολλή δουλειά τα, οι γονεί μπροστά του και πολλέ φορέ δεν έχουν το χρόνο ή τη βούληση να ασχοληθούν τόσο πολύ με τα παιδιά του. Λοιπόν, θα πρέπει να δίνονται τέτοια μαθήματα στο σχολείο και έτσι τα παιδιά να έχουν και άλλες πηγές γνώσεων για αυτά τα θέματα πέρα από το διαδίκτυο. Τα έγγραφα, τα διάφορα για την σεξουαλικοποίηση δείχνουν ότι από όταν έγινε το ίντερνετ η, βασική πηγή γνώσεων για τα παιδιά τα εκθέτει σε τέτοιες γνώσεις. Χρειάζεται σωστή ερμηνεία και σωστή εξήγηση αν εκτεθούν σε αυτές τις γνώσεις τα παιδιά. Διαφορετικά επηρεάζουν αρνητικά αυτές τις γνώσεις τη συμπεριφορά και την ανάπτυξη των παιδιών. Τα παιδιά επίσης θα πρέπει να εκπαιδεύονται ούτω ώστε να μπορούν με επιδεξιότητα να αντιμετωπίσουν τα θέματα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ξεκινήσουν διάλογο με του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, τι οργανώσει καταναλωτών, κοινωνικέ οργανώσει και οργανώσει των γονέων, ούτω ώστε να καθοριστεί το θέμα αυτό, οι συνέπειε που έχει η σεξουαλικοποίηση και πώς μπορούν να αποφευθούν οι αρνητικές συνέπειες της σεξουαλικοποίησης. Ε, οι καλές πρακτικές δείχνουν ότι αυτή η συνεργασία δεν είναι μόνο εφικτή, αλλά μπορεί να είναι αποτελεσματική και καρποφόρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα υιοθέτησε μια οδηγία για την πορνογραφία. Ε, στην έκθεσή μου αναφέρθηκα στη θέση μας όσον αφορά τη σελίδα του διαδικτύου, όπως το προμία, που προωθεί βουλημία ή ανορέξια νερβόζα, διάφορες τέτοιες διατροφικές διαταραχές. Είδα αυτή την ιστοσελίδα και είδα ότι αυτά που αναφέρονται εκεί μπορεί να είναι πολύ επιβλαβή ε, και να πειράσουν αρνητικότατα τα νέα κορίτσια. Ε, δημιουργώντας ένα κύμα διατροφικών διαταραχών, οι ψυχολόγοι συστήνουν ότι τις ιστοσελίδες θα πρέπει να υπόκεινται σε πάρα πολύ αυστηρούς ελέγχους. Αυτές οι ιστοσελίδες ίσως να ενθαρρύνουν τα νέα κορίτσια να περιορίσουν πολύ αυτά που τρώνε. Πολύ συχνά τα νέα κορίτσια πιστεύουν ότι δεν πειράζει ποια είναι τα προσόντα τους ή οι γνώσεις τους. Πιστεύουν ότι το μόνο που έχει νόημα είναι η εμφάνισή τους. Ε, και αυτό είναι ότι είναι αποφασιστικός παράγων για την καριέρα τους. Όχι τα προσόντα τους, αλλά η εμφάνισή τους, μόνο η εμφάνισή τους. Θα πρέπει στο διάλογο για τις διάφορες εμπορικές προδιαγραφές και για τις διαφημίσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτό το διάλογο. Θα είναι υποφελές κάτι τέτοιο για τα παιδιά. Οι διαφημίσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να επαναξεταστεί. Την εποχή που πολλά παιδιά βλέπουν τηλεόραση, δεν θα πρέπει να προβάλλονται διαφημίσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο. Το ίδιο ισχύει και στις διαφημίσεις στους δρόμους. Πρέπει να αλλάξουν και αυτές οι αλλαγές θα βελτιώσουν την όλη κατάσταση. Στο τέλος της εκθέσεώς μου καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθέσει μελέτες και αναλύσεις όσον αφορά την σεξουαλικοποίηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για την ώρα τα στοιχεία που διαθέτουμε είναι κατακαιρματισμένα. Η Πολωνία είναι μία από τις χώρες εκείνες που δεν τα κατάφερε δεν μπόρεσε να ερευνήσει το εύρος του φαινομένου στη χώρα μου. Κάτι άλλο που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν να διαδοθούν οι βέλτιστες πρακτικές που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τύχουν οικονομική υποστηρίξεω για να αντιμετωπίσουν αυτό το αρνητικό φαινόμενο, η σεξουαλικοποίηση των κοριτσιών αυτό το φαινόμενο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ελπίζω ότι θα με υποστηρίξετε, ότι μπορώ να βασιστώ στη συνεργασία σας. Ελπίζω να υποβάλλετε πολλές τροπολογίες που θα καταστήσουν την έκθεση αυτή ακόμα καλύτερη. Και ελπίζω αυτό το έγγραφο να μας δώσει τη δυνατότητα να καταπολεμήσουμε τη σεξουαλικοποίηση και τις αρνητικές συνέπειες που έχει με αποτελεσματικό τρόπο. Ε, νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να παρατηρηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη Βασίζομαι στη συνεργασία σας και προσβλέπω στα σχόλιά σας. Tack så för det och eh, då lämnar jag ordet fritt och eh, först går ευχαριστώ πάρα Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à féliciter Madame Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την εισηγήτρια. Δεν έχω δεν έχω διερμηνία στα πολωνικά, δυστυχώς. Dzień dobry, pani Kridlewka. Ooh, I'm impressed. <laughs> It doesn't work? Okay. It doesn't work now. Συγγνώμη. Εντάξει. Έλεγα ε, και ελπίζω να ακούτε τώρα την μετάφραση στα πολωνικά. Ήθελα να σας πω, κυρία εισηγήτρια, ότι η έκθεσή σας είναι εξαίρετη και πλήρης. Θα ήθελα να σας ε, ε, συγχαρώ γιατί αυτό το φαινόμενο της σεξουαλικοποίησης των νεαρών κοριτσιών και παιδιών είναι κάτι πολύ ε, διαδεδομένο και τώρα είναι δύσκολο να πάμε προς τα πίσω και να δούμε όλα αυτά τα φαινόμενα ε, που εμφανίζονται και επιδεινώνονται και κάνουν τα παιδιά να έρχονται σε επαφή όλο και περισσότερο με εικόνες σεξουαλικές στην τηλεόραση ή αλλού ή στο ίντερνετ φυσικά που δεν είναι ελεγχόμενο υπάρχουν εικόνες ε, που δεν είναι σωστές για τα παιδιά, ακόμα και σε κάποια περιοδικά. Αυτοί που φτιάχνουν ρούχα ε, μπαίνουν μέσα σε αυτή την τάση. Ε, υπάρχει αυτή, αυτό το πρότυπο της γυναίκας μινιατούρας, η οποία είναι πολύ διαδεδομένη και βλέπουμε ότι συνεχώς τα παιδιά εκτίθενται σε τέτοιες εικόνες που τα κάνουν να μεγαλώνουν πριν την ηλικία τους. Είναι σημαντικό λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά και να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα πλαίσιο που θα προστατέψει τα παιδιά μας. Επανέρχομαι στην παράγραφο 15 όπου μιλάτε για ε, μια συνεργασία ε, των ε, αυτών που φτιάχνουν ρούχα και πραγματικά πρέπει να εμπνευστούμε από αυτό, ε, όπως και από την ε, βιομηχανία των καλλιτικών, όπου υπήρξαν κάποιες ε, πρωτοβουλίες και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνεργασία προς κοινό συμφέρον. Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει και με τους κατασκευαστές ρούχων. Τους ενδυματολόγους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό υπάρχουν ε, άνθρωποι όπως ε, ο Καρλ Λάγκερφελτ ε, που είναι ένας μόδιστρος τον οποίο πραγματικά συχαίνομαι. Αυτός λέει ότι το 34 είναι η το small δηλαδή είναι το κατάλληλο μέγεθος για τα ρούχα. Με τέτοιες λοιπόν στάσεις και ευτυχώς δεν είναι όλοι που συμμερίζονται αυτές τις στάσεις δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι ε, προωθείται αυτό το μικρότερο μέγεθος ε, το οποίο κάνει τις νεαρές ε, γυναίκες να πέφτουν σε απόγνωση και να φτάνουν σε καταστάσεις όπως την ενοχοποίηση, την νευρική ενορεξία. Μιλάτε για τους γονείς, μιλάτε για τους διαγωνισμούς ομορφιάς στις οποίους λαμβάνουν μέρος παιδιά δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε το παιδί το οποίο ε, δεν βγαίνει πρώτο σε έναν ας πούμε διαγωνισμό και να το κάνουμε να έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που θα το οδηγήσει σε νευρική ανορεξία. Επίσης ε, πρέπει αυτό το πράγμα να το βάλουμε σε ένα ε, πλαίσιο. δεν μιλάω για απαγορεύσεις απαραίτητα, αλλά ας πούμε ένας διαγωνισμός τραγουδιού είναι σαν διαφήμιση δεν πρέπει να ενοχοποιούμε αυτού ε, που χάνουν σε τέτοιου διαγωνισμού. Υπήρχε και ένα ρεπορτάζ που μιλούσε ακριβώ για αυτή την ανόητη συμπεριφορά των γονιών, κυρίω των μητέρων που πραγματικά ενοχοποιούσαν τα παιδιά του που έρχονταν δεύτερα ή τρίτα σε τέτοιου διαγωνισμού, Μάλιστα τα τιμωρούσαν πολλέ. φορές. Εντάξει, φυσικά πρέπει να διασκεδάσουν τα παιδιά. Αυτό πρέπει να είναι ένα παιχνίδι για αυτά, όχι ένας διαγωνισμός εντάξει, να ενθαρρύνουμε την προσπάθεια μεν, αλλά να μην περνάμε και κάποια όρια. Δεν έχω και πολλές τροπολογίες ε, ε, γιατί θεωρώ ότι είναι εξαίρετη η πρότασή σας, αλλά ίσως ε, θα μπορούσαμε να πάμε και λίγο παραπέρα όσον αφορά στους κινδύνους που αφορούν στην ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών, κυρίως των νεαρών κοριτσιών, σε σχέση με αυτό το φαινόμενο το οποίο είναι ιδιαίτερα ανασυχητικό. Και ελπίζω ο Καρλ Λάγκερφελτ να, πάει να πάει στα δικαστήρια κάποια στιγμή, αυτό θα με κάνει να έχω κι εγώ μια μικρή δημοσιότητα. Συμφωνώ πλήρως μαζί σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι άκρο σημαντική έκθεση και καλύπτει ένα ευρύτατο πεδίο. Η συγκεκριά μας θέλει σε πράγματι να καλύψει πολλούς τομείς και είναι ενδιαφέρον. Θα ήθελα από την πλευρά μου να υπογραμμίσω απλά κάποιες διαπιστώσεις. Θεωρώ ότι το πιο σοβαρό είναι ότι ε, είναι επιθυμητή και ζητείται τα στις στις γυναίκες, από τα ίδια τα κορίτσια η σεξουαλικοποίηση, γιατί η κοινωνία της πρόχνει προς αυτό. Προς αυτά τα μοντέλα, αυτή τη σύγχρονη τυπολογία θα έλεγα. Cool, να είναι cool, όπως λένε και στην ηλικία τους ε, οι νέοι. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει ε, συνομιλίες ε, μικρών αγοριών ή κοριτσιών. Της ηλικίας που ανέλησε η κοριτσιων Τη ηλικία που ανελησε η συγγητρια μας. Προσπαθούν να είναι σε έξι ακόμη και αν είναι σε τρυφερή, πολύ νεαρή ηλικία. Άρα δεν έχει θέση στην ηλικιακή αυτή κατηγορία η λέξη σεξ παρά ταύτα είναι ένα όρο είναι ένα επίθετο που χρησιμοποιεί αυτή η κατηγορία. Αυτή η ηλικιακή κατηγορία. Σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια, στην παράγραφο 15, κάπου διάβασα ότι ένα από τους υπευθύνους της εταιρεία που φτιάχνουν τι κούκλε μπάρμπι έλεγε ότι ε, φτιάχνουμε μπάρμπι ακόμη και πόρνες μπάρμπι γιατί υπάρχουν πολλά είδη είναι φαύλος κύκλος. Αν η κοινωνία θέλει τέτοιου είδους ε, κούκλες για παράδειγμα και κυκλοφορούν και είναι και φτηνέ και αγοράζονται, γιατί λένε κάποιες εταιρείες που κατασκευάζουν παιχνίδια εμείς να μην κατασκευάζουμε τέτοιες κούκλες. ό,τι που λέτε είναι καλό. Εγώ αυτό το θεωρώ υπερβολικό. Υπερβολικά, υπερβολικό, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Τέλος, να πω και δύο λέξεις για την πορνογραφία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παντού στον κόσμο, ίσως, η πορνογραφία, η παιδική πορνογραφία, δηλαδή η χρησιμοποίηση παιδιών ε, για πορνογραφία είναι ένα έγκλημα. Κάποιοι όμως θεωρούν ότι είναι νόμιμη η δραστηριότητα αυτή. Είναι καλό αυτό για μας. Παραδείγματο χάρη κάποιος ψάχνει μία πορνοτενία στο Google και εμφανίζονται 5 εκατομμύρια λίματα. Αυτά μπορεί να, τα έχει, να σε αυτά να έχει πρόσβαση και κάθε παιδί. Δηλαδή δεν μπορεί να μπλοκάρει κανείς την πρόσβαση των παιδιών στο διαδίκτυο. Μπορούν να δουν ταινίε πορνό στο διαδίκτυο τα παιδιά. Έχουμε λοιπόν το θέμα της χρησιμοποίησης παιδιών στις ταινίες αυτές που είναι έγκλημα όπως είπα, αλλά έχουμε και την πορνογραφία μια ελεύθερη δραστηριότητα στο διαδίκτυο που μπορεί και έχει πολύ αρνητικέ συνέπειε αν μπορούν τα παιδιά μας να παρακολουθήσουν τέτοιε ταινίε. Θα καταθέσω κάποιε τροπολογίες να συμφωνεί η συγγήτρια και την συγχαίρω για την πολύ αυτή σημαντική της ε, έκθεση και εργασία. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Μπάστος. Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την ε, συνάδελφό μας για την εξαιρετική της έκθεση. Η πρωτοβουλία αυτή είναι πραγματικά κάτι που αποτελεί ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα και μας ε, δημιουργεί πολλές σκέψεις Υπάρχουν λοιπόν στερεότυπα τα οποία δημιουργούνται, ακόμη και στην ηλικία των 6 με 13 χρόνων. Καλή έκθεση, καλά διαρθρωμένη. Έχουμε τον ορισμό καταρχήν της ε, σεξουαλικοποίησης ε, που είναι πάρα πολύ ξεκάθαρος. Οι συστάσεις γήτρες είναι εξίσου ξεκάθαρες και από αυτόν και καθώς και ό,τι λέει η συγγήτρια για το διαδίκτυο, την τηλεόραση, για την ευαισθητοποίηση αυτών που κατασκευάζουν ε, βίντεο παιχνίδια κτλ. Δηλαδή ουσιαστικά η μεγαλύτερη ευθύνη που πρέπει να φέρουν και κάτι που ανέφερε και συνάδελφος, η μεγάλη ευθύνη της οικογένειας. Πρόκειται για ένα ανησυχητικό φαινόμενο που αυξάνεται. Και το εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να κάνει και αυτό ό,τι μπορεί για να προληφθεί ή να αποτραπεί ως το δυνατόν αυτό το φαινόμενο. Αυτή την, την ιδέα θα την προωθήσω και εγώ. Είναι καλές οι συστάσεις της εισηγήτριας, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν συστάσεις και για κάποιες ειδικέ εξτάσεις που θα πρέπει να γίνουν για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των δασκάλων που ίσως να μην έχουν υπόψη τους αυτή την άφηση του ενισχυτικού αυτού φαινομένου. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εαυτό μου. Είμαι σκιώδης για την έκθεση αυτή, σκιώδης συζητητής και νομίζω ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Εξίσου σημαντική είναι και η έκθεση και νομίζω ότι συμβαδίζει και με όσα είχαμε συζητήσει και νωρίτερα σήμερα δηλαδή για την κατάργηση ορισμένων ε, ειδών υπηρεσιών στην Ένωση και η σεξουαλικοποίηση των παιδιών σίγουρα είναι μία λυσίδα σε αυτό τον κρίκο και θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά τι είναι η σεξουαλικοποίηση. Εσείς έχετε προβάλλει διάφορες πτυχές, καλό είναι αυτό. Κάτι όμως που δεν άκουσα ή δεν είδα στην έκθεση είναι κάτι που, ναι, με το αναφέρατε εσείς, αλλά δεν έχει διατυπωθεί ξεκάθαρα στην έκθεση και είναι κάτι που μας αφορά όλους. Όταν βλέπουμε τηλεόραση, όταν παίζουμε ένα βιντεοπαιχνίδι, Εμείς μπορούμε να ελέγξουμε τι θα δει το παιδί ως κάποιο βαθμό. Όταν όμως βγει από το σπίτι και πάει στο σχολείο, υπάρχει ένα κύμα σεξουαλικό πιστό βομβαρδίζεται θα έλεγα από τη σεξουαλικοποίηση στο παιδί. Άρα είναι σημαντικό και το τι γίνεται στον έξω κόσμο, όχι μόνο στο σπίτι. Η βιομηχανία της μόδας, είπατε για το Λάγκερφελτ και το τα λοιπά. Πρέπει και αυτοί να λάβουν τις ευθύνες τους. Είναι μια πτυχή που θέλω να την ε, αναφέρετε πιο ξεκάθαρα. Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω στο σημείο 4, στην τέταρτη σύσταση δηλαδή, λέτε ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για ε, τους γονείς και τα λοιπά σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε εδώ και τα κλιπ μουσικών τραγουδιών. Έχουμε πρίες πολλές φορές σκηνέ, σκηνέ σεξ στα παιχνίδια αυτά, τα βίντεο παιχνίδια. Και όχι τόσο το τι δείχνουν, αλλά το πώς το δείχνουν. Και πάρα πολλοί κακές διαφημίσεις ε, υπάρχουν και πολύ κακά ε, κλιπ μουσικής Επίσης μίλησαμε για το διαδίκτυο, τις διάφορες ιστοσελίδες, το αναφέρατε, είναι πολύ σημαντικό, υπάρχουν πάρα πολλές ιστοσελίδες, τεράστιος αριθμός και νομίζω ότι θα ήταν καλό να μπορούμε να μπλοκάρουμε κάποιες από αυτές τις ιστοσελίδες. Δυστυχώς δεν είναι και τόσο εύκολο και το γνωρίζετε πολύ καλά γιατί είναι ένα θέμα στο οποίο πάμε έχετε εργαστεί Μπλοκάροντας ε, την ιστοσελίδα μπορεί κάποιο να μπλοκάρει και που προσπαθούν να μπλοκάρουν την ιστοσελίδα. Είναι λίγο πολύπλοκο. Μηπω θα έπρεπε να υπάρχει Παραδείγματο χάρη ε, κάποιο μηχανή που να μπλοκάρει μια ιστοσελίδα όταν ε, συναντήσει κάποιε συγκεκριμένες λέξεις. Αυτό μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, γιατί θα μπλοκάρει και ιστοσελίδε που προσπαθούν να καταπολεμήσουν την πορνογραφία στο διαδίκτυο. Αλλά περιλαμβάνω κάποιες από αυτές τις λέξεις. Πώς θα μπλοκάρουμε λοιπόν κάτι, χωρίς να υπάρχει και ασφάλεια δικαίου και χωρίς να μπλοκάρουμε και σελίδες που δεν θέλουμε να μπλοκάρουμε. Είναι λίγο λεπτό το θέμα. Τώρα, στην 7η σύσταση που έχετε διατυπώσει, δεν είμαι βέβαιος ότι καταλαβαίνω πολύ καλά ότι η σεξουαλική αγωγή θα βοηθήσει και την οικογενειακή ζωή. Θα προετοιμάσει το παιδί για την οικογενειακή ζωή. Είναι κάτι οικογενειακό. Ε, συγγνώμη, υποκειμενικό το τι είναι οικογένεια. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που εμπεριέχονται στον όρο αυτό. Γιατί μιλάμε εδώ για σεξουαλική αγωγή, για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Δεν νομίζω ότι προετοιμάζει αυτό κάποιον στην οικογενειακή ζωή και μπορεί να μην θέλει κάποιο να έχει οικογενειακή ζωή. Λοιπόν, ένα παράδειγμα ήταν αυτό. Θα σταματήσω εδώ, θα καταθέσω και εγώ κάποιε τροπολογίε και ελπίζω ότι από κοινού θα καταφέρουμε να ενισχύσουμε την ε, έκθεση αυτή. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ονομάζομαι Μάρκαρετ Τσούτ εργάζομαι στη μονάδα για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών στη Γενική Διεύθυνση Justice, δικαιοσύνη. Η Κομισιόν προ... καλωσορίζει αυτή την έκθεση. Γνωρίζουμε το θέμα της σεξουαλικοποίησης και το γεγονός ότι το φαινόμενο αυτό ε, βαίνει αυξανόμενο. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση σχετικά με το θέμα αυτό της σεξουαλικοποίησης ότι η κουλτούρα μας ε, συνεχώς περνοποιείται και γενικά νομιμοποιούνται τέτοια φαινόμενα και ούτω καθεξής. Κάποια από τα νούμερα που αναφέρθηκαν στη σχετική ακρόαση λαμβάνουν υπόψη τους, ε, για παράδειγμα, τη μουσική που ακούνε τα παιδιά το 70% των ε, τραγουδιών έχουν σεξουαλικές αναφορές. Επίσης, ε, έγινε ένα φιλτράρισμα της παγκόσμιας ε, βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών και βλέπουμε ότι έχουμε δισεκατομμύρια πορνογραφικών μηνυμάτων που μεταφέρονται μέσα από τα μέσα τηλεπικοινωνίας κάθε χρόνο. Έχουμε λοιπόν συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση ε, που είναι αρμόδια για το πιο ασφαλές ε, διαδίκτυο και να πω ότι αυτό το πρόγραμμα για το ασφαλέστερο διαδίκτυο δεν ε, περιορίζεται μόνο στον έλεγχο, γιατί δεν μπορούμε να μπλοκάρουμε και να ελέγχουμε τα πάντα. Μιλάμε περισσότερο για κατάρτιση και διαπαιδαγώγηση. όταν οι γονείς έχουν καλή επιτήρηση και έλεγχο, για παράδειγμα, όταν έχουν τον υπολογιστή στο, στην κουζίνα και βλέπουν τι βλέπει το παιδί τους, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά τώρα με το ε, ασύρματο διαδίκτυο, κανείς μπορεί να πάει στα Starbucks και να κατεβάσει ό,τι θέλει. Άρα, μεγαλύτερη έμφαση στην διαπαιδαγώγηση που θα πρέπει να δώσουμε. Στο πρόγραμμα Δάφνη του χρόνου, ε, το Δάφνη είναι το πρόγραμμα που όλοι γνωρίζετε, έχει ως στόχο την πρόληψη της βίας εναντίον των παιδιών, ε, των νεαρών ατόμων και των γυναικών μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα κάνουμε κάποια πρακτικά έργα που έχουν ε, ως στόχο τις ε, συμπεριφορικές αλλαγές ε, και τις αλλαγές τάσης και ελπίζουμε να συμπεριληφθεί κάτι μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Συνεργαζόμαστε επίσης με τους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού και Εκπαίδευσης για αυτά τα θέματα. Χαιρετίζουμε λοιπόν την έκθεση και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει κάτι επιτέλους για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σκολεύσκα. Όχι, πρώτα η κυρία Κώστα. Ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ήρθα λίγο αργά. Ζητώ συγγνώμη από την εισηγήτρια, απλώ ήθελα να τονίσω το εξή. Αυτή η έκθεση είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, με πολύ καλή διάρθρωση και φυσικά το θέμα είναι πολύ ε, ενδιαφέρον. Θα προσπαθήσω να συνεχίσω από τα σχόλια της Κομισιόν. Ζητώ από την Επιτροπή και την Εισηγήτρια να γίνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια προστασίας των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Αυτό διασυνδέεται ε, με τη συζήτηση που θα γίνει τον επόμενο Σεπτέμβριο. Με ενδιαφέρει ειδικότερα λοιπόν η δημιουργία δεσμών εδώ έτσι ώστε να ε, ασχοληθούμε με τα θέματα που αφορούν τα παιδιά, γιατί αυτά τα θέματα ε, είναι ε, θέματα που εμφανίζονται σε πολλές διαστάσεις και έχουν ενδιαφέρον για όλους μας. Να σας θυμίσω και το εξής. Υπάρχουν κάποιες γκρίζες ζώνες μεταξύ του τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο. αυτός, ε, ε, αυτό το γκρίζο πεδίο είναι πολύ ευρύ. Έτσι λοιπόν τα κράτη-μέλη και οι Κομισιόν θα μπορούσαν να προωθήσουν συμφωνίες με τους ε, χειριστές και τις εταιρείες των κινητών τηλεφώνων, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις. Ευχαριστώ. λόγω λόγος τώρα στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να ξεκινήσω Καταρχάς, να πω στην κυρία Κώστα ότι εγώ είμαι ένα πληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, αλλά με χαρά μου θα συνεργαστώ μαζί σας σε αυτό το θέμα. Αδειμονώ λοιπόν να έχουμε κάποια συνεργασία Χαιρετίζω την παρέμβασή σας και πραγματικά έχουμε μια ε, παρόμοια προσέγγιση σε αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα, το οποίο ως τώρα δεν έτυχε προσοχής. Είναι η πρώτη έκθεση για τη σεξουαλικοποίηση των νεαρών κοριτσιών. Για τον κύριο Ταραμπέλα να πω καταρχάς ότι σας ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια και για το γεγονός ότι είπατε τόσο εγκομασιατικά λόγια για την έκθεσή μου. Ε, αναφέρατε τους ε, διαγωνισμούς ομορφιάς. Είναι δύσκολο φυσικά να τους απαγορεύσουμε για διάφορους λόγους. Καταρχάς είναι μια τεράστια βιομηχανία η οποία παράγει ε, πολύ μεγάλα κέρδη για τους εμπλεκόμενους. Από την άλλη, οι γονείς έχουν κέρδος από τέτοιες ε, δραστηριότητες και πολύ συχνά θεωρούν ότι αποτελεί ε, κάτι τέτοιο ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Αν οι ίδιοι δεν έχουν επιτύχει κάτι τέτοιο, θέλουν τα παιδιά τους να το επιτύχουν. Στην Γαλλία, για παράδειγμα, υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα που ονομάζεται Mini Miss France, το οποίο, από ό,τι ξέρω, ε, διακόπηκε. Δεν αποσύρθηκε, δεν θα βγει. Γιατί η Γαλλία έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες ε, για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Ελπίζω κι άλλα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν. Ένα τώρα αυτό το σχόλιο από την πλευρά μου. Φυσικά δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε αυτούς τους διαγωνισμούς, αλλά θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να έχουμε κάποιες προϋποθέσεις. Την έγκριση του γονέα, αλλά φυσικά και την έγκριση ενός ψυχολόγου ίσως να μην αρκεί να συμφωνούν, να συνενούν οι γονείς. Θα πρέπει και ένας εκπαιδευμένος ψυχολόγος να μπορεί να, να διατυπώσει άποψη σχετικά με το αν ένα παιδί μπορεί και είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε έναν τέτοιο διαγωνισμό και να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση. Δεν έχουν όλα τα παιδιά στην ηλικία των 3 και 4 ετών το ίδιο επίπεδο ερημότητας. Θα άξιζε λοιπόν μια τέτοια προσέγγιση τώρα σχετικά με την ε, βιομηχανία του ενδύματος και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αυτές ε, οι βιομηχανίες ε, δυστυχώς, όπως σας είπα, είναι έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας και υπάρχουν λοιπόν κάποιοι περιορισμοί. Αρχικά η έκθεση μου ήταν πολύ πιο μεγάλη, αλλά οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου άμεσα παρενέβησαν και έπρεπε να κάνω πιο πυκνή την έκθεσή μου, πιο συνολική. Δεν μπόρεσα λοιπόν να δικαιώσω την προσπάθειά μου. Αναφέρω αυτό που είπε και ο Πρόεδρος. Δεν είναι όσο επαρκής και ολοκληρωμένη θα ήθελε η έκθεσή μου, αλλά δεν μπόρεσα να αλλάξω τους κανόνες. Τα φίλτρα ε, γονεϊκού ελέγχου είναι ένας τρόπος για να ελέγξουμε την πρόσβαση. Αλλά τα παιδιά σήμερα συνεχώς χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα κινητά και τα smartphones που αντικαθιστούν τα λάπτοπ και τους υπολογιστές. Αυτά είναι πέραν του ελέγχου μας οι γονείς ε, μπορεί να θεωρούν ότι αρκεί αυτό το φίλτρο του ελέγχου που έχουν τοποθετήσει στο σταθερό υπολογιστή τους στο σπίτι. Όμως δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα smartphones που προσφέρουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Έχουμε λοιπόν ένα διαβριμένο φαινόμενο, το οποίο ήθελα να αναφέρω και δεν είχα χώρο, είναι η αποστολή γυμνών και πορνογραφικών ε, φωτογραφιών μέσω του ίντερνετ. Η έκθεση δείχνει ότι το φαινόμενο της σεξουαλικοποίησης έχει καταστεί πραγματικό πρόβλημα. Όταν εγώ ήμουν παιδί η κατάσταση ήταν διαφορετική. Οι γονείς μου ήξεραν ότι δεν, δεν είχα έκθεση σε τέτοιες ε, πηγές σεξουαλικοποίησης. Σήμερα τα παιδιά έχουν έκθεση σε μεγαλύτερες τέτοιου είδους απειλές. Έχω μιλήσει με πολλές μητέρες που μου είπαν ότι είναι αβοήθητες, περιμένουν κάποια αρρωγή από τους νομοθέτες. Πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες. Πρέπει να αλλάξουν οι διατάξεις, γιατί οι γονείς χρειάζονται την υποστήριξή μας. Θα ήταν καλή ιδέα επίσης να δημιουργήσουμε μία πλατφόρμα για ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των γονέων. Για παράδειγμα, μπορεί ένας γονέας να εντοπίσει ένα παιχνίδι ηλεκτρονικό το οποίο διατίθεται και δεν θα πρέπει να διατίθεται. Να διαδώσει λοιπόν αυτή την πληροφορία στους υπόλοιπους γονείς. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ σε αυτό που είπατε σε σχέση με το άρθρο 7 και τον ορισμό της οικογένειας. Όπως το βλέπω εγώ, ε, αυτό είναι το βασικό θέμα που διακυβεύεται. Ίσως δεν έχει να κάνει τόσο με την προετοιμασία της οικογενειακής ζωής και της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Είναι περισσότερο ένας ορισμός της οικογένειας. Εκπροσωπώ εδώ την Πολωνία και στο δικό μας σύνταγμα ξεκάθαρα ορίζεται τι είναι η οικογένεια. Αυτό ήταν και το σημείο αναφοράς που χρησιμοποίησα όταν ε, ανέλαβα αυτή την έκθεση. Ταυτόχρονα κατανοώ ότι κάποιοι άλλοι δεν συμμερίζονται την άποψή μου και σέβομαι αυτή τη διαφορά άποψης. Μπορεί να έχουμε διαφορετική στάση για αυτό το θέμα. Αναγνωρίζω λοιπόν το σχολείο σας, όμως πραγματικά θα πρέπει και εσείς να καταλάβετε ότι βασίζομαι στον ορισμό της οικογένειας ως εμφανίζεται στο Σύνταγμα της Πολωνίας. Από αυτή την άποψη λοιπόν περιμένω πολλές τροπολογίες που θα βελτιώσουν την έκθεσή μου γιατί αυτή είναι η βασική μας ε, στόχευση, να έχουμε μια καλή έκθεση που θα δείχνει την πολυπλοκότητα αυτού του φαινομένου της σεξουαλικοποίησης. Ελπίζω ότι ε, οι θεσμοί μας θα συνεργαστούν με τα σχολεία και τα παιδιά έτσι ώστε τα παιδιά λιγότερο να εκτίθενται στις αρνητικές επιπτώσεις ε, της σεξουαλικοποίησης. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ε, λέγατε ότι έχουμε πρόβλημα με το κείμενο. Όμως, γνωρίζω πολύ καλά και εγώ ε, τα όρια που έχετε για το κείμενο και πολύ, πολλές φορές έχει κανείς να πει πολύ περισσότερα πράγματα αυτά που το επιτρέπει η γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλάβει σε ένα κείμενο. Έτσι έχουν τα πράγματα, έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 17 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι και 19 Σεπτεμβρίου θα γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή και τον Οκτώβριο στην Ολομέλεια. Μπορούμε να προχωρήσουμε από αυτό το σημείο και να πάμε στο σημείο 15 που αφορά το δικαιώματα και ηθαγένεια για την περίοδο 2014-2020 και δίνω το λόγο στην κυρία Μπάστος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όπως έπαιδε και από τον τίτλο, προσπαθούμε να καθορίσουμε στα πλαίσια του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου την χρηματοδότηση και την οικονομική δομή για το πρόγραμμα Δάφνη πιο συγκεκριμένα για την επόμενη αυτή περίοδο. Προσπαθήσαμε να καθορίσουμε το πολιετές πλαίσιο και να καθορίσουμε τη δομή χρηματοδότησης μειώνοντας όμως τον αριθμό των μέσων χρηματοδότησης η Επιτροπή υπέβαλε για το 2014 μέχρι το 2020 τη δημιουργία αυτού του προγράμματος για τα δικαιώματα και την ηθαγένεια, που είναι διάδοχος του προγράμματος για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ηθαγένεια, του προγράμματος Δάφνη, για την καταπολέμηση της διάκρισης και διαφορά στην προάσπιση της ισότητας ανδρών και γυναικών και διάφορα άλλα προγράμματα επίσης συμπεριλαμβάνονται όπως το Progress. Θα ήθελα να τονίσω τις εξουσίες αρμοδιότητες που έχουν διάφορες επιτροπές. Αυτό σχέδιο γνωμοδότησης καλύπτει διάφορους τομείς. Η Επιτροπή της ΛΥΜΠΕ, της Απασχόλησης και της Επιτροπής Γυναικών έχουμε όλες οι επιτροπές αρμοδιότητες σε διάφορους τομείς. Κάποιες επιτροπές είναι καθήλυνα αρμόδιες για κάποιους τομείς, Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις τρεις επιτροπές που εμπλέκονται προσπαθήσαμε να καθορίσουμε ποιες είναι οι αποκλειστικές ευθύνες και ποιες είναι οι κοινέ. Και βέβαια ε, καταλήξαμε σε αυτούς τους ορισμούς. Στη δική μας επιτροπή μπορούμε να προτείνουμε κάποιες τροπολογίες για τις εταιρεωτικές σκέψεις και τα άθρα και υπάρχουν και άλλα άλλες αιτιολογικές σκέψεις και άθρα που είναι εκτός του πεδίου μας, εκτός της εντολής μας όπως θα περιμένατε. Η βασική μας μέρημνα όσον αφορά το νέο πρόγραμμα είναι η αποφυγή της καταστάσεως κατά την οποία επιδιώκουμε πολύ αόριστους γενικούς στόχους που αφορούν την ισότητα των φίλων, ισότητα ανδρών και γυναικών και να μην πετυχαίνουμε το στόχο λόγω αοριστολογίας. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μην μειώσουμε την ορατότητα, τη σημασία του προγράμματος Δάφνη. Ούτε θα θέλαμε να αδικήσουμε το νέο πρόγραμμα για τα δικαιώματα και την ηθαγένεια. Αυτό ήταν που είχαμε υπόψη μας στην όλη προσπάθεια. Όταν συντάξαμε στην, την έκθεση που έχετε μπροστά σας. Έχω υποβάλει 18 τροπολογίες. Το πρώτο σημείο αφορά την ισότητα ε, που θα πρέπει να αναφέρεται στον ίδιο τίτλο του προγράμματος. Το πρόγραμμα θα είχε τίτλο «Δικαιώματα και ηθαγένεια». Ε, μία τροπολογία έχει υποβληθεί για να το αλλάξουμε «Δικαιώματα, ισότητα και ηθαγένεια» να γίνει ο τίτλος. 2, 3 και 6 αυτές οι τροπολογίες ενισχύουν την αρχή μη διάκρισης και τις ισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε ήταν ότι έπρεπε να διατηρήσουμε τους στόχους του παρόντος κανονισμού και του προγράμματος Δάφνη, δηλαδή καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, κάτι που ζητήσαμε στις τροπολογίες 4, 5, 15, 16 και 18. Εφόσον έχω το λόγο, θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι πρότειναν στο μέλλον να υπάρχει ένα κεφάλαιο που θα καλύπτει αυτό που συζητήσαμε, δηλαδή τη σεξουαλικοποίηση των νέων ανθρώπων. Κατά την άποψή μου είναι ζωτική σημασία η αντιμετώπιση του θέματος αυτού στην επόμενη περίοδο στα πλαίσια του προγράμματος Δικαιώματα και Ιθαγένεια και αυτό το θέμα ταιριάζει και με την άλλη φροντίδα μας για τη χρηματοδότηση που είναι η βασική μας ε, ανησυχία. Χρηματοδότηση δεν μπορεί να μειωθεί ε, περισσότερο περισσότερο από αυτό που προβλεπόταν παλιά για το πρόγραμμα Δάφνη. Εφόσον δεν έχουμε κατανοήσει, δεν γνωρίζουμε ακριβώς ε, ποιο ποσό θα διατεθεί για αυτό το πρόγραμμα, όπως βλέπουμε εμείς, εμείς, τα πράγματα, ε, εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτά που τονίσαμε στην έκθεσή μας, δηλαδή να μην μειωθεί ο προπολογισμό θα έπρεπε να παραμείνει ο προπολογισμό ως έχει, χρησιμοποιώντα την βάση του παρελθόντο. Και μάλιστα θα μπορούσε να αυξηθεί η χρηματοδότηση. στι τροπολογίε 17 και 18 ζητούμε την αναγκαία χρηματοδότηση, τουλάχιστον αντίστοιχη με τη χρηματοδότηση που είχε διατεθεί κατά το παρελθόν. Πιστεύουμε ότι αυτή η χρηματοδότηση θα αυξηθεί και δεν θα παραμείνει ως έχει. Ελπίζουμε τουλάχιστον. Και πιστεύουμε σε συνομιλίες με τους σκιώδεις εισηγητές κατέστησε σαφές ότι όλοι οι σκιώδεις εισηγητές ε, των διαφόρων ομάδων ε, υποστηρίζουν ένθερμα την μη μείωση ε, του διαθεσίμου ποσού για την περίοδο 2014-2020. Στην τροπολογία 9 διαγράφουμε την ισότητα ανδρών και γυναικών από τον κατάλογο των αρχών της μη διάκρισης και υπάρχουν δύο τροπολογίες για την πρόθεση ισότητας ανδρών και γυναικών και την καταπολέμηση της βίας κατά διαφόρων ομάδων συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Πρέπει να είναι συγκεκριμένη στόχη του προγράμματος αυτή. Θα ήθελα να υποβάλω και άλλη τροπολογία που δεν συμπεριλαμβάνεται εδώ ακόμα. Ε, θα ήθελα να συμπεριλάβω και τη βία κατά των ηλικιωμένων. Και ένα άλλο σημείο το οποίο θα ήθελα να προσεγγίσω και να αναφέρω είναι ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αναφέρεται αυτό στις τροπολογίες 12 και 16. Και τέλος, οι 13 και 17 υπογραμμίζουν τη σημασία της τακτικής συλλογής συγκρίσιμων στοιχείων όσον αφορά τις διάφορες μορφές βίας. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αν με επιτρέπετε, θα ήθελα να αναφερθώ στο όλο χρονοδιάγραμμα και την προθεσμία για τις τροπολογίες που παρετάθη μέχρι 17 Ιουλίου 12 το μεσημέρι. Οι τροπολογίες θα συζητηθούν στις 13 Δεκεμβρίου και στις 20 Δεκεμβρίου θα ληφθεί απόφαση και περιμένω οι ασδήποτε τυχόν συνεισφορές έχετε. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, πάρα πολύ. Η ε, κυρία Κροστέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ήταν πολύ χρήσιμο αυτό που, η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε μεταξύ μας και με τους Κιώδης για την προετοιμασία της ε, συνεδριάς, λέει κύριε Κώστα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία αυτή που θίξατε. Δηλαδή που θα πρέπει να μπει η λέξη ισότητα στον τίτλο, συμφωνώ να διευρυνθεί ο τίτλος. Ανησυχώ λίγο όμως, διότι αυτά τα προγράμματα, τα συγχωνευόμενα, που μπαίνουν στον πολιτή προγραμματισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάποιες περιπτώσεις δι... ίσως μπορεί να ενσωματώσουν διάφορες πτυχές και έτσι να μην είναι αναγνωρίσιμα πλέον αυτά τα προγράμματα, να μην είναι αναγνωρίσιμοι οι στόχοι, κάποιοι στόχοι που για μας είναι απόλυτα ε, υποστηρίξιμοι. Εγώ θα έλεγα ότι η σύσταση που έκανε το Κοινοβούλιο και που επανέλαβε και στην τροπολογία 4 η κυρία Λεμπάστος ε, είναι να κρατήσουμε αυτούς τους στόχους την καταπολέμηση κατά των διαφόρων μορφών βίας, όχι μόνο κατά των γυναικών, αλλά και των ανηλίκων και των εφήβων. Αυτό αφορά το πρόγραμμα Δάφνη και αυτό θα πρέπει να το προασπιστούμε. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν θα είναι δυνατόν. Θα πρότεινα το εξή να διατηρήσουμε τουλάχιστον τον υπότιτο Δάφνη. Είναι να χάσουμε μια, ένα σήμα, μια μάρκα σαν το Δάφνη θα ήταν σφάλμα και εκτός του πλαισίου να πω κάτι, τη συζητήσεων, ξέρουμε πόσο τα brand είναι επενδύσεις. Αυτές, η, ο τίτλος μιας εταιρεία. Χρησιμοποιούν εταιρείε πάρα πολλά χρήματα επί σειρά ετών να δημιουργήσουν αυτή τη φήμη, το όνομα. Το να χάσουμε λοιπόν αυτή την αφορά, αυτό το brand, αυτό το τίτλο, αυτή τη μάρκα είναι παρακινδυνευμένο. Ε, ε, λοιπόν, ε, δεν βρήκα κάποιον που να συμφωνεί ε, με να μην υπάρχει αυτή την αναφορά. Λοιπόν, θα κάνω τέτοια τροπολογία σχετική. Ελπίζω να γίνει αποδεκτή αυτή η τροπολογία και από τη συναδελφό Μπάστο και από του άλλου συναδέλφου και από την συγκίτρια Γκόντ. Αλλά γνωρίζω ότι σίγουρα είναι διθέσιμο το δεκτή αυτό που λέω. Δεύτερον, αριθεύει ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίω επί των, γυναι... των θεμάτων για τι γυναίκε και για του ανήλικου και για τι εφήβου. Σαν Επιτροπή Γυναικών, σω θα ήταν χρήσιμο όμω να αναφερθούμε και σε κάποιες άλλες τυπολογίες μορφές διάκρισης και βίας και σε άλλα πλαίσια από την οπτική, τη γυναικεία οπτική γωνία όσον αφορά τα διάφορα στερεότυπα, την εικόνα των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης ε, όσον αφορά το θέμα της υποστήριξης των διαφόρων ενώσεων και των υπηρεσιών και των δράσεων και των προγραμμάτων που θέλουν να επανεντάξουν γυναίκες ε, μετά το εμπόριο λευκής σαρκός, παραδείγματος χάρη, ή τα παιδιά, ή τα άτομα που έχουν υποστεί κάθε μορφή βίας, υπό διάφορες μορφές λοιπόν, πιστεύω και χρειάζονται μορφές υποστήριξης για τα διάφορα είδη παρέμβασης που θα μπορούσαν να προταθούν. Οι βέλτες πρακτικές για την πρόληψη της βίας και υπό τη μορφή συμβουλών προς τα βία άτομα Έχουμε πολύ, ε, σε διάφορε χώρε έχουμε γίνει διάφορε δοκιμέ πολύ ενδιαφέρουσε. Θα πρέπει να γίνεται παρέμβαση και προ αυτή την κατεύθυνση. Όχι μόνο όσον αφορά το θύμα, αλλά όσον αφορά και τον θήτη. Ε, λοιπόν, θα κάνω σχετικέ τροπολογίε, θα υποβάλω. Συγχαρητήρια για την κυρία Μπάστο, γιατί η έκθεσή τη είναι μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο για μια κομφάρα στον εαυτό μου διότι είμαι σκηγόντης εισηγητής και για αυτό το θέμα. Έτσι έχουν τα πράγματα να κάνουν. Συμφωνώ με όσα είπαν οι κυρία Κώστα και Μπάστος. Πράγματι είχαμε πρόσφατα μια συνεδρίαση για τις τροπολογίες, η οποία διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και χαίρομαι πολύ που έγιναν αυτές οι προτάσεις, γιατί νομίζω ότι ενισχύουν το ποιοτικό σκέλος. Την ποιότητα της πρότασης, τροπολογίες 9, 10, 11 και 12, χαίρομαι που κατατέθηκαν και είναι πολύ καλές τροπολογίες. Χθε συζητήσαμε επίσης κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ή βελτίωσης του κειμένου. Όμως, από ό,τι φαίνεται, η πρότασή μας πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες όπως εμείς τις αντιλαμβανόμαστε. Και αυτό είναι το κατώτατο που μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή δεν μπορεί η χρηματοδότηση να πέσει κάτω από αυτό το όριο που έχουμε. Αυτό πρέπει να γίνει αποδεκτό. Θα πρέπει επίσης να πούμε, μάλιστα, ότι θα πρέπει και να αυξηθεί. Όχι από αυστηρά οικονομική σκοπιά, αλλά έχοντας υπόψη μας την κοινωνία. γιατί όλα αυτά κοστίζουν και θα πρέπει να δούμε πού εντοπίζονται οι ανάγκες της κοινωνίας. Θα πρέπει να κάνει η Επιτροπή μας και τους σχετικούς υπολογισμούς. Εμείς λέμε ότι υπάρχει ανάγκη να διατεθούν περισσότεροι πόροι σε αυτό το πρόγραμμα. Εάν τώρα αργότερα προκύψει μια διαφορετική εκτίμηση, θα δούμε πώς θα το χειριστούμε, αλλά σε αυτή τη φάση Νομίζω ότι πρέπει να εμείνουμε στη θέση μας. Κάτι άλλο σημαντικό, το ανέφερε η κυρία Κώστα. Εγώ θα έλεγα ότι το Δάφνη και οι πόροι που έχουν προβλεφθεί για αυτό το πρόγραμμα να διατηρηθούν και κυριότερο να μείνει το σήμα αν θέλετε Δάφνη. Δεν ξέρω αν αλλάξει κάποια στιγμή το όνομα του προγράμματος, αλλά το Δάφνη έχει κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να διατηρηθούν. Μπορεί να του βάλουμε έναν υπότιτλο, δεν ξέρω. Θα πρέπει να δούμε τι προτάσεις μπορούμε να διατυπώσουμε σχετικά. Ώστε νεολογικά να κρατήσουμε το Δάφνη έχει. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ. Οπότε με αυτά και με αυτά νομίζω ότι τώρα μπορούμε να δώσουμε το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, καλωσορίζουμε τη γνωμοδότηση. Συγχαίρουμε την εισηγήτρια, είναι πολύ καλά συνταγμένη η έκθεση. Όπως είπε και η εισηγήτρια, αυτό το πρόγραμμα για τα δικαιώματα και την ηθαγένεια έχουν να κάνουν και με, με δύο σκέλη του Progress και με το Δάφνη. Στόχος μας είναι η, γνωμο... η χρηματοδότηση των προγραμμάτων να διατηρηθεί. Ιδίω δεν να μείνει η χρηματοδότηση στο τομέα τη ισότητα ανθρώπων και γυναικών και για την ε, χρηματοδότηση του Δάφνη. Στόχος μας ήταν να υπάρχει απλούστευση με βάση και την συνολικότερη πρόταση για το πολιτές μουσονομικό πλαίσιο. Καλωσορίζουμε τις προτάσεις που περιλαμβάνει η γνωμοδότηση και τις αλλαγές που προτείνονται. Οι στόχοι και οι προθέσεις αναφέρονται απλά πιο αναλυτικά. Ε, πάντως τις έχουμε ήδη και εμείς ως Κομισιόν εκφράσει. Για, την, για τον προπολογισμό να πω ότι το ποσό που θα τεθεί στο πρόγραμμα δεν θα αποφασιστεί από το ίδιο το πρόγραμμα. Εμπίπτει στι διαπραγματεύσει για το πακέτο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Άρα, πιθανέ αλλαγέ ή σχετικέ διαπραγματεύσει είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο μια διαφορετική διαδικασία. Επίση, το πρόγραμμα δικαιοσύνη που προτείνει γραμματικά Justice, δικαιοσύνη, θα προέβλεπε την συμπληρωματικότητα, ιδίως σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων σε ποινικέ ε, διαδικασίε. Και το τελευταίο έχει να κάνει με τον ε, προγραμματισμό και το χρονοδιάγραμμα. Θέλω να τονίσω ότι ο προγραμματισμός για την έγκριση θα πρέπει να είναι στο δυνατόν πιο σύντομα να ολοκληρωθεί για να μπορέσουμε να περάσουμε στην υλοποίηση Θα εκτιμήσουμε λοιπόν ε, την ταχεία δεκπαιρέωση του θέματος από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μπάστος έχει τώρα το λόγο για να συνοψίσει, να κλείσουμε με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ και τη Σίλβια Κώστα ε, αναφέρθηκε σε αυτά που συμφωνήσαμε όσον αφορά τις ανησυχίες που αφορούν όλες τις πολιτικές ομάδες. Ανησυχίες που σχετίζονται με τον τίτλο, τη μάρκα, ούτως η Δάφνη. Κυρίως όσον αφορά την ε, αποτίμηση του προγράμματος Δάφνη, θα ήταν καλό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κρατήσει τη μάρκα, το όνομα Δάφνη που χρειάστηκε πολλές επενδύσεις στο Δάφνη και πολλές προσπάθειες. Αυτή η μάρκα λοιπόν δεν θα πρέπει να μείνει στο περιθώριο. Θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στο ευρύτερο πρόγραμμα όσον αφορά την ηθαγένεια, τα δικαιώματα και την ισότητα. Η ιδέα που υπευλήθη να παραμείνει σαν υπότιτλος το Δάφνη. Είναι μια λογική πρόταση και πραγματικά καλύπτει τις ανησυχίες που εκφραζόταν για τη συνεχιζόμενη ορατότητα του προγράμματος Δάφνη και την εκμετάλλευση της επιτυχίας που είχε το πρόγραμμα Δάφνη από τη δεκαετία του 90. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε, θα πιέσουμε και ελπίζουμε ότι θα υποβληθούν σχετικές τροπολογίες όσον αφορά την χρηματοδότηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ενστερνίστηκε το στόχο μας. Δεν θα θέλαμε η χρηματοδότηση να είναι χαμηλότερη από, αυτό που, από το ποσό που είχε διατεθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και θα πρέπει βεβαίως να λάβουμε υπόψη τα όσα συμβαίνουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Με βάση αυτό το υπόβαθρο αυτό το κονδύλι του προϋπολογισμού θα μπορούσε και να αυξηθεί και αρκετά. Είναι θέμα κοινή λογικής. Αν περνά κανείς μια οικονομική και κοινωνική κρίση όπως είναι η παρούσα, αυτό που τίνει να συμβεί είναι ο κόσμος να ασκεί περισσότερη, μεγαλύτερη ψυχολογική και σωματική βία κατά των πλέον ευαλώτων, όπως είναι οι γυναίκες και τα παιδιά. Αυτό είναι ένα αυξανόμενο φαινόμενο στα πλαίσια της κρίσης. Θα πρέπει να αντιδράσουμε λοιπόν, να ανασκουμπωθούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα για την πρόληψη, πρόληψη που είναι ένας βασικός άξονας του προγράμματος. Μπορεί να υπάρχει χρήσιμη επικάλυψη αυτού του προγράμματος με το πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη, το Justice. Ας μην το λησμονούμε αυτό όταν θέλουμε να αυξήσουμε τον προπολογισμό. Περιμένω ανυπόμονα να δω τις τροπολογίες που θα υποβάλουν οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Äh, Να σας πω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για την έκθεση Μπάστος είναι 17 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Και θα ξανασυζητήσουμε στις 3 Σεπτεμβρίου και η Επιτροπή θα ψηφίσει στις 19 έως 20 Σεπτεμβρίου. Με αυτό μπορούμε τώρα να τελειώσουμε με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Τώρα πάμε στο σημείο 16. Πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία παθήσεων των γυναικών. Για να είμαστε ξεκάθαροι γι' αυτό, σε περίπτωση που δεν έχετε πάρει αυτό το έγγραφο στη γλώσσα σας, θα μεταφραστεί σε κάθε γλώσσα, αλλά αυτή τη στιγμή το έχουμε μόνο στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά. Μόλις ε, έχουμε διαθέσιμη τη μετάφραση, θα σας την δώσουμε και σε περίπτωση που το θέλετε ε, και δεν είναι στη γλώσσα σας διαθέσιμο, θα το έχετε τότε. Ας δώσουμε τώρα το λόγο στην συγκίτρια την κυρία Τζελίλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να καθησυχάσω τους συναδέλφους σε λίγο θα είναι διαθέσιμες όλες οι γλωσσικές εκδοχές και η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι το Σεπτέμβριο. Άρα υπάρχει άπλετος χρόνος ε, για να λυθεί το κείμενο. Να γίνουν όλες οι διορθώσεις και οι βελτιώσεις. Σκοπός της ε, εκθέσεως είναι να επικεντρωθούμε επί της προλήψεως των ασθενειών των γυναικών, ασθενειών που συνδέονται με την ηλικία, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έτους της ενεργού, της δραστήριας γύρανσης και της αλληλεγγύης των γενεών. Όπως σημειώθηκε αυτό το ευρωπαϊκό έτος που είναι αφιερωμένο στην ε, δραστήρια γύρανση, στην ενεργό γύρανση, και πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια αυτού του έτους ήταν σημαντικό να αφιερώσουμε ε, μια αναφορά στις γυναίκες ιδιαίτερη και να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα επειδή βλέποντας τα στατιστικά στοιχεία βλέπουμε ότι το φάσμα του ευρωπαϊκού πληθυσμού που είναι πάνω από τα 65 από 87 εκατομμύρια ανθρώπους έχει περίπου 51 εκατομμύρια γυναίκες. Άρα το ποσοστό του πληθυσμού πάνω από τα 65 απαρτίζεται ε, κυρίως από γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι έχουν προσδόκιμο ζωής μεγαλύτερο. Και αυτό είναι καλό, αλλά όλα τα στατιστικά στοιχεία μας λένε ότι τα χρόνια τα παραπάνω που ζουν οι γυναίκες, κανονικά αυτά τα χρόνια, κατά μέσο όρο, τα ζουν σε συνθήκες που δεν είναι ιδιαίτερα θετικές, αυτό διότι οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από τη φτώχεια για πολλούς παράγοντες. Διότι δεν έχουν ίσως εργαστεί πάντα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Διότι η ανεργία πλήττει περισσότερο τις γυναίκες από τους άντρες. Επειδή οι γυναίκες πολύ συχνά κάνουν δουλειές που δεν είναι τυπικές, διότι πληρώνονται λιγότερο. Οπότε σωρεύουν και λιγότερες συνταξιδοτικές εισφορές. Λοιπόν, οι ηλικιωμένε γυναίκες γι' αυτό έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν στη φτώχεια. Ε, επίσης, μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και μοναξιάς, διότι πολλές γυναίκες ζουν μόνες τους. Ε, καταλήγουν να ζουν μόνες τους. Οι γυναίκες μετά, σε αυτά τα χρόνια που ζουν περισσότερα, υπόκειται σε ασθένειες και πολύ σοβαρές ε, που οδηγούν σε αναπηρίες ε, ε, όπως η νόσος του Αλσχάιμερ. Όλες οι νευρο, νευρικές, νευροεκφυλιστικές ασθένειες που είναι το περισσότερο τις γυναίκες από τους άντρες και υπάρχουν και άλλες ασθένειες, σειρά ασθενειών που πλήττουν τις γυναίκες όπως οι καρδιαγγειακές ασθένειες που εσφαλμένως θεωρούνται πρόβλημα τυπικά, των, τυπικό των ανδρών. Πράγματι οι άντρες ε, πλήττονται περισσότερο από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι γυναίκες λιγότερο, να μόνο μέχρι μια κάποια ηλικία. Μετά τα 45-50 οι γυναίκες ε, ε, κινδυνεύουν εξίσου όπως και οι από αυτές τις ασθένειες. Μετά υπάρχουν και άλλες ασθένειες που αφορούν τις γυναίκες, συντυπικές των γυναικών, αυτές που συνδέονται με μυοσκελετικές ασθένειες. Άρα είναι καλό να αναπτυχθεί μια στρατηγική πρόληψη η οποία να αφορά όλος ιδιαίτερος τις γυναίκες. Αυτό αυτό, γι' αυτό αξίζει τον κόπο να επενθυμίσουμε και την επιστημονική έρευνα, τη φαρμακολογική έρευνα που ε, γίνεται κυρίως βασικά επί των ανδρών και αυτό είναι σφάλμα διότι διάφορες παθολογίες, διάφορες παθήσεις ή ε, καρδιαγκιακές εκδηλώνονται επί των γυναικών με έναν τρόπο διαφορετικό ε, σε σύγκριση με τους άντρες και τα συμπτώματα είναι διαφορετικά η διάγνωση ή φάρμακα που γίνονται βάσει πειραμάτων εντό εισαγωγικών επί των ανδρών σημαίνει ότι δεν προλαμβάνονται επακριβώς και σωστά οι ίδιες ασθένειες ε, όταν πλήττουν τις γυναίκες. Ε, κλείνω λέγοντας και ελπίζω ότι οι συνάδελφοι θα μπορέσουν να διαβάσουν ε, τη δική μου πρόταση, το κείμενό μου, αλλά βεβαίω θα είμαι ευτυχής να εμπλουτίσω το κείμενό μου με πολλές συνεισφορές. Και θα θυμίσω λοιπόν ότι ο στόχος είναι αυτός, είναι ο εξή. Να συμμετάσχουν οι εθνικές αρχές, οι τοπικές αρχές στην προσπάθεια της πρόληψης που εδράζεται πολύ επί της ενημέρωσης. Ενημέρωση λοιπόν καλύτερη, πιο διάχυτη, δεδομένη, πιο λεπτομερής που θα μπορέσει να βοηθήσει τις γυναίκες που ζουν περισσότερο, να ζουν όμως και πολύ καλύτερα. Και συνεπώς να ξεπεράσουμε το ευρωπαϊκό έτος για την ε, ενεργό γύρανση, την δραστήρια γύρανση. Να είναι ένα έτος αφιερωμένο σε αυτά τα προβλήματα, αλλά και στην πραγματικότητα τα κράτη-μέλη θα πρέπει σε συνεργασία προφανώς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαμορφώσουν προγράμματα και στρατηγικές για την πρόληψη και την ενημέρωση και βοήθεια όσον αφορά τα προβλήματα αυτά για τις γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Τζιλίλη Μπορεί να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση με την κυρία Τσόβη στον πρώτο, να έχει το πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. δεδομένου ότι φέτος το έτος έχει ανακηρυχθεί ως ε, το έτος της ενεργούς συγκύρανσης και δεδομένης της σημασίας αυτού του θέματος είναι απαραίτητο να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και να επικεντρωθούμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις ε, ασθένειες των γυναικών που σχετίζονται με τη γύρανση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ε, να έχουμε αυτή την έκθεση η οποία είναι ιδιαίτερα αντικειμενική. Όμως θα πρέπει να την βελτιώσουμε περαιτέρω. Για παράδειγμα, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε όλες τις γυναίκες που ζουν μόνες τους, δηλαδή αυτές που πάσχουν από τη μοναξιά. Μόλις χθες το απόγευμα είχαμε την Ιταλική έκδοση της έκθεσης και σήμερα την Αγγλική. Δεν την έχω στη γλώσσα μου την έκθεση. Θα ήθελα να διαβάσω όλη την έκθεση, ούτως ή άλλως όμως ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε ως τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. κυρία Παλιαδέλη. Ε, να ευχαριστήσω καταρχήν την συνάδελφο, την κυρία Αντζελίλη, για την πρωτοβουλία με αφορμή το έτος ενεργού γύρανσης ε, να περιλάβει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά την, ε, τις αρρώστιες που σχετίζονται με τις γυναίκες και τον τρόπο που αντιμετωπίζονται. Αναρωτιέμαι βεβαίως, και αυτό είναι μια ερώτηση, αν η ένταξη της πρωτοβουλίας, της πρότασης αυτής στο έτος της ενεργού γύραρσης απαγορεύει να συμπεριληφθούν στο κείμενό σας, στο κείμενο της ε, αναφοράς, ε, της έκθεσης ε, και τροπολογίες που σε ένα βαθμό τις βλέπω εδώ μέσα έχουν σχέση όχι αναγκαστικά με την ηλικία αλλά έχουν σχέση με τις γυναίκες. Ένα παράδειγμα είναι ότι ενώ αναφέρονται στοιχεία από το Διεθνές ε, Ινστιτούτο για την έρευνα του καρκίνου αναφέρεται ως ε, μία από τις δυνατότητες πρόκλησης ε, η μαστογραφία για τον καρκίνο του μαστού φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αναφερθεί και το, τεστ, το PAP test για την έρευνα, για, τον εντοπισμό του καρκίνου της μήτρας για παράδειγμα που είναι εξίσου είναι κατεξοχήν γυναικεία γυναικείος καρκίνος, αποκλειστικά γυναικείος καρκίνος. Ε, που αυτό όμως δεν περιορίζεται μόνο στις ηλικιωμένε γυναίκες, αλλά ε, εκτείνεται στο, σε όλο τον εύρος ηλικιών του γυναικείου φύλου. Επομένως, εκτιμώ ότι ανεξάρτητα από το αν η έκθεση σχετίζεται κυρίως με τις μεγαλύτερες ηλικία γυναίκες, δεν μπορούμε να περιλάβουμε μέσα σε, αυτά, μέσα σε αυτήν και προτάσεις οι οποίες στις οποίες ε, στηρίζεται η μελλοντική υγεία των γυναικών ακόμη κι αν εντοπίζεται η ασθένεια νωρίτερα. Το ίδιο ισχύει, ε, η ίδια παρατήρηση νομίζω ότι έχει σχέση και με τις ορμόνες που είναι επίσης ένα και τις επιπτώσεις τους με τις αλλαγές που προκύπτουν στο γυναικείο φύλλο μετά από ορισμένε ε, περιόδους, δηλαδή στην έναρξη της ορμονικής δράσης και στην πάυση της ορμονικής δράσης και σε ασθένειε που σχετίζονται με αυτέ, ανεξάρτητα από την ηλικία. Επομένω, η ορμονική ε, εξέταση των γυναικών ανεξαρτήτως της ηλικία μπορεί να προλάβει όπως και ο διαβήτης πράγματα που μπορεί να προκύψουν στην επόμενη ηλικία, στις μεγαλύτερες ηλικίε. Επομένως ε, θα έλεγα ότι θα πρέπει να, αλλά εδώ θέλω τη γνώμη της ε, εισηγήτριας, με αυτή την αφορμή να ζητήσουμε από την Επιτροπή να διευρύνει την ενημέρωση και να απαιτήσει έρευνες ε, που δεν έχουν σχέση μόνο με τις γυναίκες μιας συγκεκριμένης ηλικία και πέρα, αλλά έρευνες οι οποίες θα βοηθήσουν τις γυναίκες να ενημερωθούν σωστά και τους γιατρούς να εξειδικευτούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν γυναικείες ασθένειες, ασθένειες με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωποι το γυναικείο φύλλο και που εμφανίζονται κάποια ώριμη στιγμή της ζωής τους, αλλά όχι αναγκαστικά. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον ε, ότι δεν έχουμε εξειδικευμένες περιπτώσεις διάγνωσης διαφορετικών εκδηλώσεων ασθενειών όπως είναι το μυοκάρδιο, η, η, του μυοκαρδίου και ότι επομένως δεν υπάρχουν γιατροί πολλοί που θα μπορούσαν να εντοπίσουν τις διαφορετικές εκδηλώσεις αυτής της ασθένειας στις γυναίκες και να μην τις μπερδεύουν με τις ανδικές. Λοιπόν, και προς αυτή την κατεύθυνση και χαίρομαι ότι το επισημαίνετε, νομίζω ότι πρέπει ε, να, να, προχωρήσουμε και να το ε, εντείνουμε, να την ε, πίεσή μας. Και πραγματικά πιστεύω όλο, ότι έτσι κι αλλιώς η γεροντολογία που είναι ένας κλάδος όχι ιδιαίτερα διαδεδομένος στις χώρες της Ευρώπης ότι θα έπρεπε να ενθαρρυνθούν και τα πανεπιστήμια και τα εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα να, ε, να, επιβάλλουν την ανάπτυξη αυτής της ειδίκευση, η οποία δεν αφορά μόνο τις γυναίκες αλλά μπορεί να εξειδικευτεί και στις γυναίκες. Επομένως η γεροντολογία είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει πολύ την ε, ε, Ευρώπη και με αφορμή το έτος γύρανσης, της ενεργού γύρανσης, αλλά γενικότερα και ως εξειδίκευση στο γυναικείο φύλλο ειδικότερα. Ε, έχουμε το χρόνο να κάνουμε και ε, συζήτηση και περισσότερες τροπολογίες με την ε, έκθεση αυτή, την οποία θεωρώ πολύ σημαντική και με αφορμή την ενεργό, το έτος για την ενεργό γύρωση, αλλά και ως ερέθισμα για την εξειδίκευση και των ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιστημονικών κέντρων προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ επομένω πολύ την εισηγήτρια ε, για την πρωτοβουλία αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Tack det och då går ordet till fru Merci, monsieur le président. Deux sujets. Κύριε Πρόεδρε, Καταρχάς, ε, να ξεκινήσω λέγοντας πως αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα προσπαθήσω και εγώ να καταθέσω τροπολογίες σε δύο συστάσεις. Καταρχάς, ε, θα θεωρώ ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις ε, γυναίκες που ζουν στις αγροτικές περιοχές που έχουν ακόμα πιο πολύπλοκα προβλήματα από ότι γενικώ οι ηλικιωμένε γυναίκες. Για παράδειγμα, στη χώρα μου, που είναι η Ρουμανία, έχουμε ένα πραγματικό ε, πρόβλημα με τους ε, γιατρούς που φεύγουν από τη χώρα και πηγαίνουν αλλού να δουλέψουν. Υπάρχουν λοιπόν νοσοκομεία στα χωριά μας που κλείνουν. Υπάρχουν ε, πολύ λίγοι εξειδικευμένοι γιατροί. Και έτσι οι γυναίκες οι ηλικιωμένες στις αγροτικές περιοχές είναι ακόμα πιο δύσκολα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον θα πρότεινα τα κράτη-μέλη και οι Κομισιόν να ενθαρρύνουν τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις να κάνουν εκστρατείες που ε, θα ασχοληθούν με τα πολύ σοβαρά προβλήματα της ε, γύρανσης. Ας πούμε, προγράμματα ευαισθητοποίησης των γυναικών να τις οδηγούν στο να πάνε στο γιατρό και στο νοσοκομείο. Δυστυχώς λόγω της κρίσης υπάρχουν λίγα χρήματα για κάτι τέτοιο. Όσον αφορά σε προγράμματα δηλαδή που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση. Υπάρχουν λοιπόν πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες ε, θα μπορούσαν ε, να μπουν σε αυτό το πεδίο των εκστρατιών ε, και των ερευνών γιατί θα ήταν κάτι πολύ χρήσιμο να υπάρχει λοιπόν ενθάρρυνση των εθελοντών να κάνουν τέτοια πράγματα σε αυτόν τον πολύ σημαντικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο, η εκπρόσωπος της Κομισιόν, κυρία Ντελαμάτου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ήταν στα Ιταλικά και μπορέσαμε να τη διαβάσουμε και να ετοιμάσουμε την απάντησή μας. Καταρχάς, ε, χαιρόμαστε που η έκθεση ευθυγραμμίζεται με την εργασία που κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει μια διαδικασία διαβούλευσης για τις ε, χρόνιες ασθένειες. Σε αυτή τη διαδικασία ε, δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη προσέγγιση στο φύλλο, αλλά γενικά μιλάμε για τις ε, ασθένειες λόγω γύρανσης. Μιλήσατε για το καρκίνο, τις καρδιακές νόσους, το διαβήτη. Θεωρούμε ότι είναι ξεκάθαρο πως κάποιες νόσοι πλήττουν διαφορετικά τις γυναίκες από τους άντρες. Διαφορετικά είναι τα συμπτώματα και δεν γνωρίζουν πάντοτε οι επαγγελματίε στον χώρο της υγείας αυτά τα στοιχεία. Εργαζόμαστε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι είναι μια εξαίρετη ευκαιρία ε, οι χρόνιες νόση, τα χρόνια νοσήματα να ε, αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης. Υπάρχει και άλλη μια διαδικασία που είναι μια στρατηγική για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών που έχουν συγκεκριμένη αναφορά στην υγεία, συγκεκριμένα δηλαδή στις διαφορές ε, που έχουν τα δύο φύλλα σε θέματα υγείας. Υπάρχουν σεμινάρια ευαισθητοποίησης ε, στα κράτη-μέλη που μιλούν για αυτές τις διαφορές ε, των προβλημάτων υγείας στις γυναίκες και στους άντρες. Έγινε ένα τέτοιο σεμινάριο και νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως είπα όλοι όσοι ασχολούνται με τις γυναίκες και τους άντρες δεν γνωρίζουν πάντοτε τις διαφορές σε αυτά τα προβλήματα υγείας. Δεν μιλάω για τα νούμερα, αλλά για τα ειδικά συμπτώματα και τις θεραπείες. Ακόμα και στη φαρμακευτική βιομηχανία πραγματικά φαίνεται ότι κάποια φάρμακα ε, δεν αντιμετωπίζουν ε, με τον ίδιο τρόπο την νόσο όταν είναι σε άντρα και όταν είναι σε γυναίκα. Στην έκθεσή σας αναφέρεστε σε πολλά θέματα. Μιλάτε για το κάπνισμα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια καμπάνια, μια εκστρατεία για το υπερβολικό κάπνισμα για τις γυναίκες, όχι μόνο για τους ε, ηλικιωμένους, όπως ανέφερε κάποιος άλλος ευρωβουλευτής. Μιλάμε για την συλλογή δεδομένων επίσης. Εμείς συνεργαζόμαστε με τη Eurostat ε, για να ασχοληθούμε με το θέμα της συλλογής δεδομένων αναφύλο. Έχουμε τους δείκτες εκεί. Θέλουμε να βελτιωθεί η ποιότητά του στα κράτη-μέλη και επίσης συνεργαζόμαστε με άλλους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με τη συλλογή δεδομένων, τον ΠΟΗ και τον ΟΑΣΑ, για να βελτιωθεί η ποιότητα με το στόχο να έχουμε τα ίδια στοιχεία, τα ίδια δεδομένα και να έχουμε γρήγορα διαθέσιμα τα δεδομένα. Για παράδειγμα, κάποια ε, δεδομένα για την θνησιμότητα ε, είναι για το 2009 και καλό θα ήταν να έχουμε περισσότερα στοιχεία και άλλα που να σχετίζονται με την νοσηρότητα, γιατί όταν έχουμε προγράμματα πρόληψης πρέπει να γνωρίζουμε πώς έχει η κατάσταση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον λοιπόν είναι να εξετάσουμε όλα τα στοιχεία, τα στοιχεία που αναφέρετε στην εκθεσή σας και γενικά να πω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε γιατί συνάδουν αυτά που προτείνετε με αυτά που ήδη κάνουμε. Ευχαριστώ λοιπόν για την έκθεση, για τις τροπολογίες που θα ενδεχομένω θα καταθέσετε και για να σας δώσουμε κάθε βοήθεια που μπορεί να χρειαστείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κώστα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να εκφράσω βεβαίω την ικανοποίησή μου για αυτή την έκθεση προ τη συνάδελφα Αντζαλίλη, διότι πρόκειται περί θέματο επί το οποίο είναι σωστό το Κοινοβούλιο να διερωτηθεί περισσότερο και να επεξεργαστεί και κάποιες συστάσεις. Μεταξύ άλλων αυτό είναι ένα έτος που μπορεί να θέσει στο προσκήνιο αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να επενθυμίσω τρία θέματα που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά συμμεριζόμενοι ουσιαστικά τα σημεία που ήδη θίγησαν. Το πρώτο είναι το εξή. Το θέμα που η παραπομπή στο πρόγραμμα Horizon, το πρόγραμμα έρευνα, που είναι πολύ σωστό. Το έθιξε η εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μια δράση θετική που νομίζω ε, είχαμε βάλει μια γυναίκα όταν ήμουν επίτροπος για ισότητα που ήταν ειδική επί, ε, φαρμακολόγος στην Επιτροπή την Ενιαία για το Φάρμακο. Μια επιτροπή που σε κάθε κράτος ε, μέλος υπάρχει και καθορίζει αυτή η επιτροπή και ετοιμάζει και στα, πώς γίνονται οι στατιστικές και έρευνες. Η συμμετοχή της ήταν συμβολική. Πολύ συχνά εκεί όμως ε, δεν γίνεται αξιολόγηση της διαφορετικές συνέπειες που έχει η έρευνα και τα φάρμακα και οι θεραπείες και η συμπταμοντολογία ε, που είναι διαφορετική για τις γυναίκες από ό,τι για τους άντρες. Ε, ε, και επίση λαμβάνοντα υπόψη και το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωή για τι γυναίκε. Το άλλο που είναι σημαντικό είναι η έρευνα, όπω έλεγε η κυρία Παλιαδέλη, να είναι πιο εστιασμένη. Γίνονται πολλέ προ... για την πρόληψη. Στη χώρα μου και όχι μόνο, οι γυναίκε έχουν γίνει πιο πολύ καπνίστριε από του άντρε, κυρίω οι νέε γενιέ των κοριτσιών. Έχουμε καθησυχάσει πολύ και στι χώρε και σε Ευρώπη όσον αφορά τις ζημιές που κάνει το αλκοόλ και ο καπνός. Έχουμε, είμαστε πρώτη θέση δυστυχώς στην Ιταλία. Οι Ιταλίδες γυναίκες είναι οι μεγαλύτερες καπνίστες στην Ευρώπη. Και οι νέοι της Ιταλίας που πριν, μέχρι πριν από 10 χρόνια δεν έπιναν πολύ, τώρα έχουν την τάση να γίνονται αλκοολικοί. Εμείς είχαμε επικρίνει αυτή την έλλειψη προσοχής σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα ε, για την ε, νέα γενιά, διότι έχουμε καθησυχάσει πιστεύω. Ε, και όσον αφορά και τους θανάτους κλπ. Και αυτά στην προχωρημένη ηλικία δημιουργούν πολύ μεγάλες ζημιάς. Μετά έχουμε την κατάθλιψη και τη μοναξιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεται στην έκθεση, που γίνεται μια αναφορά στα φάρμακα που παίρνουν οι ηλικιωμένε κατά της κατάθλιψης. Χρειάζεται όμως να υπάρξει και μία μορφή ε, πρόληψης, που ίσως φαίνεται να απόμακρη, αλλά όπου έγινε ήταν σημαντική. Πρέπει να προσφέρουμε στις γυναίκες της τρίτης ηλικίας ή στις τέταρτης ηλικίας δυνατότητες πολιτισμικές, εκπαιδευτικές. Υπάρχει με τα πανεπιστήμια της ηλικίας που είναι διαδομένο πείραμα σε όλη την Ιταλία και εκεί 75% είναι γυναίκες που πηγαίνουν. Εκεί είναι μια δεύτερη ευκαιρία, second chance, για κοινωνική επαφή και έχουν θεραπευτικό αποτέλεσμα. Πρόσφατα είχαμε στατιστικά στοιχεία στην Ευρώπη που έδειχναν πως το να συμμετέχει κανείς σε μορφές πολιτισμικής δραστηριότητα έχει πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα στην υγεία και πολύ συχνά ψυχοσωματικό το αποτέλεσμα. Και δίπλα από αυτό ε, και άλλες παρέμβασεις μπορούν να γίνουν. Η βοήθεια στην κατοικία είναι πάρα πολύ, πρέπει να συσταθεί πολύ ε, όσον αφορά σε σύγκριση με την νοσοκομιακή περίθαλψη και η προσφυγή σε νέες μορφές ε, ιατρικής και να παρακολουθούμε και ποια είναι η κατάσταση των μοναχικών ατόμων και σε μικρά κέντρα κλπ. Οι ηλικιωμένε γυναίκες είναι αυτές που περιθάλπουν, caregivers. Και εκείνες ακόμα και όταν έχουν δυσκολίες οι ίδιες, προβλήματα υγείας, πολύ συχνά θεραπεύουν τι επόμενε γενιέ. προσέχουν. Είναι κάπως γυναίκες σάντουιτ, αν θέλετε, πρέπει να το προσέξουμε. Η ηλικιωμένη γυναίκα που παρόλο που έχει ε, προβλήματα υγεία με τη σειρά τη είναι υπεύθυνη για άλλα άτομα, για άλλα πρόσωπα. Όχι μόνο ο σύζυγος, μπορούν να άλλα πρόσωπα τη οικογένεια με διάφορα προβλήματα. Άρα θα πρέπει να ε, δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε αυτόν τον πυρήνα ε, που έχουν αυτές οι γυναίκες και ανθρώπους που εξαρτώνται από αυτούς. Ε, ε, υπάρχουν πολλές γυναίκες σε αυτήν την κατάσταση. Ε, θα ήθελα να πω στον πρόεδρο, στον άντρα πρόεδρο, που είναι ευαίσθητος με τα θέματα, σας το λέω σε εσά κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας πω ότι ξέρω ότι πολύ συχνά οι άντρες ηρωνεύονται και λένε ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο παρόλο που λέμε ε, αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσα να πω ότι ένα επιχείρημα υπέρ της θεραπείας για τους άντρες και τις γυναίκες πρέπει να συμφιλειωθούν περισσότερο, όταν συμφιλειώνται περισσότερο οι ρόλοι κάνει κανεί να ζει περισσότερο, αυτό πρέπει να πούμε. Όταν μιλάμε πολύ για το γεγονός ότι πρέπει να δίνουμε περισσότερη προσοχή στην πολιτική της συμφιλίωσης, οι γυναίκες έχουν πολύ περισσότερους ρόλους και ίσως αυτό παίζει ρόλο και ζούμε περισσότερο. Ε, το σκέφτομαι, προβληματίζομαι από αυτού. Διότι φαίνεται να ταιριάζει με τα στοιχεία που συζητούμε όσον αφορά τι διάφορε παθολογίε που εμφανίζουν στι γυναίκε. Ευχαριστώ πολύ. Να υπογραμμίσω αυτό που είπατε στο τέλο. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άντρε που κοροϊδεύουν και κάνουν αστεία για το γεγονός οι γυναίκες ζουν περισσότερο. Συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν έχει μόνο να κάνει με την εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των γυναικών, αλλά και των αντρών. Ο λόγος ε, είναι τώρα στην κυρία Αντζελίλη, την εισηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ξέρω ότι ασχολείται πάρα πολύ μαζί με την Ευρωστάτ προσπαθώντας να συλλέξει και να επεξεργαστεί μετά τα στοιχεία με τον πιο επικαιροποιημένο και τον πιο χρήσιμο τρόπο. Ακόμα και αν γνωρίζω ότι η Ευρωστάτ, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητούν από τα κράτη-μέλη μεγαλύτερες προσπάθειες για τη συλλογή στοιχείων, πιο συγκεκριμένων στοιχείων και συνεπώς πλέον χρησίμων στοιχείων. Ευχαριστώ μετά όλες τις συναδέλφους που πήραν το λόγο και τις διαβεβαιώ για μία ακόμη φορά ότι σύντομα θα έχετε το κείμενο σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές και υπάρχει και χρόνος για να ε, υποβληθούν διάφορες τροπολογίες, να εμπλουτίσουμε το κείμενο, να εμβαθύνουμε στο θέμα. Θα ήθελα να πω από τώρα ότι συμφωνώ με όλες τις παρατηρήσεις οι οποίες ακούστηκαν και επί της ιδέας, της προτεραιότητας να επενδύσουμε στην πρόληψη κατά τη διάρκεια όλης της φάσης του κύκλου ζωής, διότι η πρόληψη πρέπει να γίνεται από όταν είμαστε μικροί. Παιδιά, ναι, είναι θέμα εκπαίδευσης για τη σωστή υγεία, για την πρόληψη των ασθενειών, που προφανώς ε, συμπεριλαμβάνει επίσης και καλή εκπαίδευση όσον αφορά τη διατροφή, καλή διατροφική παιδεία, ε, για την κατανάλωση κυρίως την κατάχρηση του αλκοόλ, του, του, του φαγητού επίσης, υπερβολικό φαγητό και το κάπνισμα. Πρόληψη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής είναι το κλειδί, ούτω ώστε μετά να έχει κανείς μια τρίτη ηλικία σε καλή, με καλή υγεία. Και αυτό ισχύει και για τις ε, νευροεκφυλιστικές ασθένειες που αφορούν τον εγκέφαλο, διότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι ασθένειες εκφυλιστικές που ίσως ε, προέρχονται από διάφορες πηγές. Ε, συμφωνώ να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες στην Ήπεθρο, διότι σαφώς ε, βρίσκονται σε συνθήκες ιδιαίτερης μοναξιάς, ιδιαίτερων δυσκολιών όσον αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις πληροφορίες. Όσον αφορά τώρα τις πληροφορίες, αληθεύει ότι περνάμε μια περίοδο κρίσης, οπότε δαπανώνται λιγότερα χρήματα και για την πρόληψη και ακόμα λιγότερα χρήματα για την ενημέρωση. Διότι οι πληροφορίες θεωρούνται ίσως, πώς να το πω, κάτι παραπάνω, περιτό και όχι υπερτεραιότητα Θα ήθελα να προσθέσω και παραθέτω τον εαυτό μου σαν παράδειγμα. Ήθελα να πω λοιπόν ότι παρά το ότι μπορεί να είναι κανείς πολύ καλά εκπαιδευμένος, που είμαι πολύ προσεκτική με αυτά που συμβαίνουν και ζω, πώς να το πω, σε διεθνέ, διεθνείς συνθήκες, πρόσβαση σε πάρα πολλές πληροφορίες. Εγώ ίδια όμως ήμουν θύμα μια σειράς ε, προκαταλήψεων, ε, κακής ενημέρωσης, κακών πληροφοριών. Παράδειγμα, όλη η πρόληψη που αφορά την περίοδο της εμεινόπαυσης, που πολύ συχνά ε, θεωρείται σαν ένα είδος παθολογίας. Μία περίοδος παθολογική θεωρείται και πώς να το πω, περάσματος από τη νέα ηλικία, τη γόνιμη ηλικία, καλής υγείας, προς την ηλικία, πώς να το πω, σχεδόν γύρανσης. Με τη χειρότερη έννοια του όρου δεν είναι πλέον γόνιμη ηλικία, οι γυναίκες κατά κάποιο τρόπο συνοδεύονται προς μια κατάσταση, πώς να το πω, προς ένα ρόλο δευτερεύοντα. Επ' αυτού θα ήθελα να προβληματιστώ, γιατί πολλοί ψυχολόγοι μου πρότειναν να κάνω αυτή την παρατήρηση, ότι πολλές γυναίκες καταχρώνται την αισθητική χειρουργική, διότι είναι ένας τρόπος για να αισθανθούν ξανά νέες, σε μια κοινωνία που επιβάλλει μοντέλα ε, νεότητας, ε, αποτελεσματικότητας. Όμως, αντίθετα, μια, μια γυναίκα αν συνοδευτεί με έναν τρόπο υγιή να αντιμετωπίσει μια φάση της ζωής, δραστήρια ενεργή, το δει θετικά, όπως έλεγε η κυρία Κώστα, με μια ένταξη κοινωνική, με πολιτισμικές δραστηριότητες, κοινωνικές δραστηριότητες και ενδεχομένως ε, να μπει και σε κάποιο κύκλο κατάρτισης και έγινε ένα, το το έκανε ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που λέει ότι πολλά άτομα που ξεπερνούν τα 65 έτη στην ηλικία θα ήθελαν είτε να απολαύσουν τη σύνταξη, να μην εργαστούν σε πλήρη απασχόληση, full time, αλλά να εργαστούν λίγο όμως να εργαστούν σε διάφορες μορφές για να αισθάνονται ότι είναι ακόμα δραστήριοι αυτοί οι άνθρωποι και ότι ε, ε, είναι εντός της κοινωνίας και είναι χρήσιμοι. Και ίσως, όχι είπες, υπενθύμιζε η Σίλβια, όχι απλώς, ε, πώς να το πω, σαν άτομα που ίσως μπορούν να δώσουν και μια δουλειά αυτά τα άτομα και στο σπίτι δωρεάν, όχι μόνο να εργάζονται δωρεάν, να δίνουν βοήθεια στα μέλη της οικογένειας και θεραπεία που αυτή η δουλειά ε, δεν είναι πάντα θετική. Εντάξει, είναι κάτι θετικό στο σωστό βαθμό, αλλά όταν γίνεται αυτό μια δουλειά που απορροφά όλο το χρόνο και γίνεται εκμετάλλευση εντός του πυρήνα της οικογένειας, σίγουρα δεν είναι κάτι θετικό. Ευχαριστώ λοιπόν ε, όλους τους συναδέλφους οι οποίοι ε, είπαν αυτά που είπαν, ε, κράτησα πολλές σημειώσεις. Καλό μέσω τροπολογίες να εμπλουτίσουν το κείμενο το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα, παρουσίασα ένα πρωτόλιο αν θέλετε, το οποίο χρειάζεται να εμπλουτιστεί. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω τώρα για το χρονοδιάγραμμα, για την έκθεση αυτή. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 10 Σεπτεμβρίου. Το είπε σωστά και η κυρία Αντζελίλη. Η Επιτροπή μας θα ψηφίσει για την έκθεση αυτή στις 10 Οκτωβρίου. Και το Δεκέμβριο του 2012 η έκθεση θα πάει στην Ολομέλεια. Ολοκληρώνουμε λοιπόν και ερχόμαστε στο σημείο 17 που είναι η συνεδρίαση των συντονιστών που θα γίνει σε λίγο και 18 είναι η η ε, ημερομηνία της επόμενη συνεδρίασης. Δεν έχουμε τα συντονιστές ούτε τίποτε άλλο. Να σας πω πριν πότε είναι η επόμενη συνεδρίαση, πότε θα είναι. Να πω ήταν πολύ μεγάλη τιμή, μεγάλο προνόμιο που ε, συμμετείχα σε αυτήν την επιτροπή με τόσο αφοσιωμένα μέλη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πολιτικούς συμβούλους στη Γραμματεία, οι οποίοι κάνουν τεράστια δουλειά για όλους μας. Και τέλος να ευχαριστήσω όλους τους διερμηνείς που μας βοήθησαν να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε. Διότι είναι καταπληκτικό το ότι κάθομαι εγώ και σας μιλώ ειδικά και με καταλαβαίνετε. Για να δώσω το λόγο στην κυρία Οβή. Τι είπατε, έχω μια ερώτηση. Οι τροπολογίες είπατε, η προθεσμία είναι 10 Οκτωβρίου ή 10 Σεπτεμβρίου. 10 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, ωραία. Πρόεδρος. Φαντάζομαι ότι και εσείς, ε, όπως και εγώ, ανυπομονείτε πλέον για τις διακοπές. Και σας εύχομαι να έχετε όλοι σας καταπληκτικές καλοκαιρινές διακοπές. 3 Σεπτεμβρίου θα τα ξαναπούμε. 3 με 6.30. Γεια σας.